Ε, που παρακολουθεί ε, τους προπολογισμού των κρατών μελών. Ε, στο μέλλον κανένα κράτος δεν θα μπορεί να παραβιάζει τα κριτήρια αυτά. Ευχαριστώ πολύ.